So, schönen guten Morgen. Darf ich alle bitten, Platz zu nehmen? Παρακαλώ πάρτε Καλημέρα σε όλους. Και καλώ ορίσατε σήμερα λοιπόν στη σημερινή μας συνεδρίαση η πρώτη τελευταία κατά πάσα πιθανότητα τη επιτροπή Απασχόλησης για την τρέχουσα θητεία. Είναι σύντομη σχετικά η σημερινή ημερήσια διάταξη. Και αντίθετα με το σχέδιο που έχετε στην ε, διάθεσή σας, έχουμε και κάποιες αλλαγές. Έχουμε την έγκριση των πρακτικών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, Στη συνέχεια έχουμε τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία στην ημερήσια διάταξη. Μάλλον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και μετά ευρωπαϊκές στατιστικές. Αυτά για την ημερήσια διάταξη. Και έχουμε προβλέψει και μία οικογενειακή φωτογραφία. Να μην το κάνουμε αυτό στην αρχή να το κάνουμε στο τέλος της συνεδρίασης για να έχουμε όσο πιο πολλούς μπορούμε μαζί μας. Μετά την ε, ψηφοφορία νομίζω ότι θα ήταν η πιο δέουσα στιγμή. Ich muss Okay, alles klar. So, dann darf ich recht Να καλωσορίσω στην αίθουσά μας ε, και μια ομάδα επισκεπτών από την Ούνα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιανού επισκέπτες. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην πρώτη τελευταία μας συνεδρίαση. Έχουμε λοιπόν τώρα τα πρακτικά. 18 Μαρτίου 2019. Έχετε μήπω ε, καμία αντίρρηση, κάποια παρατηρήση να κάνετε, αν όχι, εγκρίνονται τα πρακτικά. Έχουμε λοιπόν τώρα το σύστημα, το συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης. Προβλεπόταν ψηφοφορία η οποία και δεν μπορεί να λάβει χώρα. γιατί έχουμε διαπραγματεύσει των σκιωδών και το Συμβούλιο ακύρωσε την δική του ψηφοφορία, άρα ούτε εμείς θα ψηφίσουμε σήμερα. Χρειάζονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Αλλά η Jean Lambert ζήτησε να πάρει το λόγο για να τοποθετηθεί. Εν συντομία. Όχι, Jean, δεν θέλεις το λόγο. Εντάξει. Όχι, λοιπόν, δεν θέλει το λόγο η Jean Lambert. Ευχαριστώ πολύ. Άρα διεκπαιρεώθηκε το θέμα αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε και στην επόμενη συνεδρίαση θα σας κάνουμε μία ενημέρωση για το πώς προχωρούν τα πράγματα. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό θέμα στην τρέχουσα θητεία. Και έτσι λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 5 της μερικής διάταξης, ευρωπαϊκές στατιστικές. Εδώ έχουμε ψηφοφορία, η οποία και θα λάβει χώρα ηλεκτρονικά. Μία και μόνη ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές, λέει ο πρόεδρος. Ψηφίστε παρακαλώ. Υπέρ κατά, ό,τι και να ψηφίσετε, ψηφίστε. Ui, 41 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, εγκρίνεται λοιπόν το κείμενο και να δώσουμε συγχαρητήρια στον εισηγητή τον Τάμας Μεσρίτς, ο οποίος δυστυχώς σήμερα δεν μπορεί να παραβρεθεί. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν την ημερήσια διαταξή. Και πρωτού πάμε στην οικογενειακή ε, φωτογραφία, γιατί ήταν και η πιο σύντομη συνεδρίαση όλων των εποχών. Πρωτού Πάμε να βγάλουμε τη φωτογραφία λοιπόν. Η επόμενη συνεδρίαση είναι 14 και 15 στο Στρασβούργο. Στην οποία περίπτωση θα πρέπει να αποφασίσουμε για τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά σας παρακαλώ τώρα για να μαζευτούμε όλοι εδώ μπροστά να βγάλουμε αυτή την επωνομαζόμενη οικογενειακή φωτογραφία εδώ ψηλά.